Το λόγο έχει εκ μέρους του Συμβουλίου ο εκπρόσωπος της Ολλανδικής ε, Προεδρίας, Χανής ε, Πλεσά. Και κυρία Χανής Πλεσά, εμείς ε, νιώθουμε ιδιαίτερο σεβασμό για σας που εκπροσωπείτε σήμερα το Συμβούλιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Mr. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ημερομηνία αυτή, 23 Ιανουαρίου του 2016, θα περάσει στην ιστορία σαν μια ιδιαίτερη στιγμή στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Οι περισσότεροι πολίτες της ε, Μεγάλης Βρετανίας αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σεβόμαστε την απόφαση αυτή και θλιβόμαστε βαθιά συγχρόνως. Όμως πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει ενότητα στον τρόπο με τον οποίο απαντάμε στο γεγονός αυτό. Σήμερα λοιπόν εκπροσωπώ εδώ ολόκληρο το Συμβούλιο, το δηλαδή και τις 28 χώρες μέλη και θα το κάνω αυτό όσο παραμένει το Ενωμένο Βασίλειο μέλος του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, είναι ένα αξιοσέβαστο μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1973 και συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα και τα άλλα ε, κράτη-μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί μια ευημερούσα και ασφαλής Ευρώπη. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος βέβαια είναι μια βασική στιγμή στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστορία όμω και η γεωγραφία δεν αλλάζουν. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι και πάντα θα είναι μια, ένα ευρωπαϊκό έθνος συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες, ε, έχουμε τις ίδιες ελπίδες και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας ως ε, εταίροι. Με άλλα λόγια, είναι προς το συμφέρον όλων μας να διασφαλίσουμε ότι μια μελλοντική σχέση θα είναι επικοδομητική και αμοιβαία θα υποφελεί και τις δύο πλευρές. Να είμαστε ξεκάθαροι. Κανείς, κανείς δεν πρόκειται να υποφεληθεί αν κρατήσει πάρα πολύ αυτή η αστάθεια. Σίγουρα το μπαλάκι είναι στο γήπεδο του Ηνωμένου Βασιλείου και περιμένουμε τα νέα του Λονδίνου σύντομα. Συγχρόνως όμως, ας δώσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να πάρει κάποιες αποστάσεις, να πάρει τις σωστές αποφάσεις και να δει πώς θα προχωρήσει. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι δηλαδή λοιπόν. Από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1957 έχει προχωρήσει και έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Έχει τη μεγαλύτερη περίοδο ειρήνης, ενοποίησε την Ευρώπη. Ήταν η ηγετική δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να κρατήσει όλο τον κόσμο ενωμένο μέσα στους κόλπους της και περισσότερο ισχυρό. Ποτέ δεν είχαμε τόσο πολύ ελευθερία τόση ευημερία και τόση σταθερότητα στην Ευρώπη. Ποτέ άλλοτε όσο σήμερα. Στην Ουκρανία ο κόσμος θυσιάζεται για να προσεγγίσει στην Ευρώπη. Γιατί, Γιατί οι άνθρωποι στην Αφρική, στην Ασία εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους, τις χώρες τους για να φτάσουν στις δικές μας ακτές. Αυτό γίνεται εξαιτία των θεμελιωδών αξιών που είναι κοινέ μεταξύ μας. Των θεμελιωδών ελευθεριών από τις οποίες εμπνεόμαστε. Αν κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Θα βρούμε το δρόμο μας. Τα επιτεύγματα αυτά, λοιπόν, είναι πραγματικά και είμαστε περήφανοι που συνεισφέραμε σε αυτά. Τίποτα όμως δεν είναι σίγουρο και τίποτα δεν είναι αναπόφευκτο. Το σοκ αυτό του δημοψηφίσματος πρέπει να μας κάνει όλους να ξυπνήσουμε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, τα αισθήματα ε, μεγάλης μερίδας του βρετανικού λαού υπάρχουν και αλλού, σε άλλε χώρε μέλη. Συνεπώ πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε τι προσπάθειές μα. Πρέπει να έχουμε μια αποτελεσματική, μια πιο αποδοτική και πάνω απ' όλα μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να πείθει περισσότερο. Τώρα εντελώ ξεκάθαρα. Στον κόσμο αυτό που ζούμε σήμερα, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες εντάσεις. Ναι, πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας. Να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό να δίνουμε τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες μας. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν η οποία θα κρατήσει τη γραμμή της. Όμως θέλουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην τη βλέπει κανείς σαν απειλή στην εθνική ταυτότητα, αλλά σαν επέκταση της δικιάς μας εθνικής ταυτότητας. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην τη βλέπει κανείς σαν ένα γραφειοκρατικό σώμα, αλλά κάποιον που διευκολύνει τις διαδικασίες. Ούτε η Ευρώπη όμως το σύνολό της, αλλά ούτε και καμία χώρα μέλος από μόνη της ή έθνος από μόνο του δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του απομονωμένο. Γι' αυτό και πρέπει να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, τις προσπάθειές μας, ώστε αυτή η ειρήνη και η σταθερότητα που έχουμε πετύχει όλες αυτές τις δεκαετίες να συνεχιστεί. Και μόνο τους αυτούς μας θα έχουμε να κατηγορήσουμε αν δεν τα καταφέρουμε. Πρόεδρε, χρειαζόμαστε την ενότητα γιατί οι πολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις γύρω από την Ευρώπη θα συνεχιστούν και πιθανόν θα πολλαπλασιαστούν. Χρειαζόμαστε την ενότητα γιατί κανείς δεν θα διστάσει να μας επιτεθεί. Χρειαζόμαστε την, ε, την ενότητα για να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ουρές, ε, ροές οι οποίες φτάνουν στις ακτές μας. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές από μόνη της. Είναι περίπλοκα όλα αυτά. Οι προκλήσεις αγνοούν τα σύνορα. Πρέπει λοιπόν να πιστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι η ενότητα είναι η καλύτερη επιλογή. Τα λόγια όμως, τα ωραία τα συμπεράσματα, οι δηλώσεις δεν φτάνουν. Πρέπει να δράσουμε. Το γεγονός ότι ο κατακαιρματισμός δεν είναι κάτι αδιανόητο, πρέπει να μας ταρακουνήσει όλους και να μας αναγκάσει να προχωρήσουμε σε δράση. Φυσικά δεν λέω ότι πρέπει να είμαστε μυρολάτρες, παραμένουμε ισχυροί. Είμαστε εκείνοι που υποστηρίζουν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο το κράτος δικαίου, την ελευθερία, τη δημοκρατία και μια οικονομία που να βασίζεται στην αγορά. Αλλά θα ήταν ανόητο να υποτιμήσουμε τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Πρόεδρε, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αυτού μας άφησε με μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο πολλοί στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αλλού νιώθουν αβέβαιοι για τις συνέπειες. Έτσι λοιπόν είναι προς το συμφέρον όλων μας να υπάρξει σαφήνεια για το τι θα γίνει στη συνέχεια και αυτό πολύ σύντομα. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι υπάρχουν οι κανόνες για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση συντεταγμένα. Όπως γνωρίζετε υπάρχει το άρθρο 50 της συνθήκης που προβλέπει τη διαδικασία εφόσον μια χώρα μέλος αποφασίσει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αρχίσει σιγά σιγά τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι στο χέρι της Βρετανική κυβέρνηση και κανενός άλλου να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 και οι διαπραγματεύσεις μπορούν να αρχίσουν μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η κοινοποίηση αυτή. Συγχρόνω, βέβαια, μένουν και άλλα να κάνουμε. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο στον Ηνωμένο Βασίλειο δεν σημαίνει ότι οι απειλέ και οι προκλήσει μα, οι κοινέ απειλέ και προκλήσει έχουν εξαφανιστεί. Ούτε σημαίνει ότι το κάθε έθνο θα τα καταφέρει καλύτερα να δράσει μόνο του, αντί να δράσουμε συλλογικά. Αντίθετα θα έλεγα. Συνεπώ, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει πράγματι να φύγει, τότε η Ένωση των 27 θα συνεχίσει μαζί μπορούμε και θα αντιμετωπίσουμε τις κοινέ προκλήσεις προκειμένου να πετύχουμε ανάπτυξη, ευημερία και ένα ασφαλές περιβάλλον που θα προστατεύει τους πολίτες μας. Αυτό ακριβώς προσδοκούν και από εμά οι πολίτες και σωστά. Η θεσμική συζήτηση για αλλαγές στη συνθήκη σίγουρα είναι ο παράδεισος των δικηγόρων και των διπλωματών. Πρέπει όμως να γίνονται για να βοηθήσουμε τους πολίτες. Συνεπώς πρέπει να ανασκουμποθούμε και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Χωρίς καμιά αμφιβολία δεν θα είναι πάντα εύκολο να συμφωνήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Είναι μεγάλη πρόκληση να λειτουργήσει η συνεργασία. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, θέτουμε σε κίνδυνο την ευημερία των λαών μας. Και αυτό, Πρόεδρε, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Συνεπώ, σε λίγε ώρε θα συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να προκαταλάβω τι συζητήσει που θα γίνουν εκεί, ούτε μπορώ να περάσω σε λεπτομέρειε για τα επόμενα βήματα. Αυτό όμω που μπορώ να κάνω είναι να σα πω ότι θα ακούσω τη συζήτησή σα προσεκτικά. Εσεί, Πρόεδρε Σούλ, θα απευθυνθείτε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα το απόγευμα και θα μεταφέρετε το περιεχόμενο του ψηφίσματος που θα εγκρίνεται σε λίγο εδώ σε αυτό το σώμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου και τώρα έχει το λόγο ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούμκα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Προεδρεύουσα, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Το Ευρωκοινοβούλιο ετοιμάζεται να συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα το πρωί είχα πολλά ραντεβού, αλλά αποφάσισα να έρθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η θέση μου σήμερα, αυτή τη στιγμή, είναι εδώ, nos ε, amis ε, Οι Βρετανοί φίλοι μας εκφράστηκαν με καθολική ψηφοφορία και είναι σαφές ότι η έκφραση της ε, λαϊκής βούλησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους. Πρόκειται για τη δημοκρατία και οφείλουμε να σεβαστούμε τη Βρετανική δημοκρατία. Και οφείλουμε να σεβαστούμε την έκφραση της βούλησης του Βρετανικού λαού. Είναι η τελευταία φορά που χειροκροτείτε εδώ. Και μάλιστα εκπλήσαμε που είσαστε και εδώ. Εσείς δώσατε μάχη για να φύγετε. Οι Βρετανοί σας ακολούθησαν. Γιατί είσαστε εδώ σήμερα. Εκφράστηκε λοιπόν ο Βρετανικό λαό με καθολική ψηφοφορία και πρέπει να σεβαστούμε αυτή την έκφραση. Δεν τολμώ να πω ότι είμαι φίλο τη Δημοκρατία για να μην αποδείξετε ότι δεν είμαι. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε την επιλογή των Βρετανών πολιτών. Εκφράστηκαν και επομένω θα πρέπει να υπάρξουν και συνέπειε. Ζητώ λοιπόν μια διευκρίνηση, όχι άμεση, γιατί το βρετανικό σύστημα είναι πιο περίπλοκο από ό,τι φανταζόμασταν. Ψηφίστηκε κάτι, αλλά υπάρχουν α, δισταγμοί. Ο κύριος Χίλο, μου, δέχεται αυτές τις συνέπειες. Διάβασα διάφορα, άκουσα διάφορα, ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ότι οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, σχεδόν όλων εκτός από κάποιες, αντέδρασαν συναισθηματικά στα αποτελέσματα της Βρετανικής ψήφου. Η Ευρώπη δεν είναι μια κεφαλική ιστορία μόνο. Φυσικά θα πρέπει να σκεφτούμε με το κεφάλι μας, αλλά όταν αισθανόμαστε θλιμμένοι πρέπει να μπορούμε να το λέμε. Και εγώ είμαι θλιμμένος μετά από αυτή την ε, ψήφο. Και δεν το κρύβω. Δεν θέλω να πέσω σε συναισθηματισμούς. Είναι βαθιά μου πεποίθηση. Πίστευα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παραμείνει στο πλευρό μας για πάντα αλλά αποφάσισε διαφορετικά και θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Ζητώ λοιπόν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και θα δω σήμερα πιο αργά τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου γιατί και ο Βρετανικός λαός παραμένει φίλος μας παρά την ψηφοφορία και το αποτέλεσμα. Θα του ζητήσω λοιπόν να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν την κατάσταση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να παραταθεί αυτή η αβεβαιότητα. Λέω λοιπόν ότι είμαι θλιμμένο. Παρότι γενικά στην πολιτική ζωή δεν μας αρέσουν τα συναισθήματα. Το λέω όμως γιατί δεν είμαι ρομπότ. Δεν είμαι τεχνοκράτης, γραφειοκράτης. Δεν είμαι γραφειοκράτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκλέχθηκε από αυτήν εδώ την σύνοδο, από αυτή τη συνέλευση, μέσω μιας ε, δημοκρατικής διαδικασίας. Είμαι εδώ σαν άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή, δεν είμαι ρομπότ, είμαι Ευρωπαίος και έχω το δικαίωμα να πω την άποψή μου για την Βρετανική ψήφο. Και να πω ότι λυπάμαι για αυτήν. Θα ήθελα το Ηνωμένο Βασίλειο να διευκρινίσει τη θέση του. Όχι σήμερα, όχι αύριο το πρωί σε 9, αλλά γρήγορα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να παραταθεί αυτή η αβεβαιότητα. Εγώ αντίθετα από άλλους δεν είμαι σκλάβος των χρηματαγορών, αλλά παρατηρώ την αντίδρασή τους. Εσείς είστε, εγώ δεν είμαι. αλλά είναι μία ένδειξη μιας γενικής κατάστασης, ε, ενός γενικού συναισθήματος. Θα ήθελα το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπα, να διευκρινίσει τη θέση του. Δεν θα ήθελα αυτή η εντύπωση να υπάρξει ότι θα γίνουν μυστικές διαπραγματεύσεις και κλεισμένων των θυρών μεταξύ των εκπροσώπων του Ηνωμένου Βασιλείου, των εθνικών κυβερνήσεων, των επιτρόπων και των γενικών διευθυντών απαγόρευσα στους επιτρόπους να συζητήσουν με τους εκπροσώπους των Βρετανών, είτε αυτών που ήταν υπέρ της εξόδου, είτε υπέρ της παραμονής. Απαγόρευσα, παρότι δεν είναι το σύστημά μου αυτό. Τους είπα δεν θέλω τέτοιες συζητήσεις. Όχι κοινοποίησεις, όχι διαπραγματεύσεις. χάσαμε. Μετά από αυτή την Βρετανική ψήφο, μία πτέρυγά μας. Υπάρχει η πτέρυγα των ιδρυτικών κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα από του άλλου. Ξεκίνησαν τη διαδικασία, αλλά δεν είναι οι μόνοι οι οποίοι την προωθούν. Και τα νέα κράτη-μέλη, όπω τα λέμε, είναι και αυτά κράτη-μέλη 100%. Εγώ χαιρετίζω την επανένωση της Ευρώπης, την συμφιλίωση και χαιρετίζω και τα νέα κράτη-μέλη. Και τα καλωσορίζω. Η Βρετανική ψήφος απέκοψε μία πλευρά μας. Μία φτερούγα μας. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να πετάμε. Θα πετάμε προς τους ε, μελλοντικού ορίζοντες της Ευρώπης και του πλανήτη. Αυτοί που μας παρατηρούν από μακριά ανησυχούν, πρέπει να το ξέρετε. Άκουσα και είδα διαφόρους ηθήνοντες, ξένους, είναι πολύ ανήσυχοι, γιατί ανησυχούν για την πορεία που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως θα πρέπει να, καθησυχάσουμε και τους Ευρωπαίους και αυτούς που μας παρατηρούν από πιο μακριά. Συνεχίζει η πτήση η πτήση αυτή έχει συγκεκριμένο στόχο. Δεν γίνεται τυχαία. Το καθορίζουν οι συνθήκες και η θέληση πολλών Ευρωπαίων. Συνεχίζει αυτή η πτήση. Και παρότι μας έχει φρενάρει λιγάκι η Βρετανική ψήφος, θα πρέπει να προοδεύσουμε προς τους στόχους που είναι κοινοί, με μια νέα αναζωογονημένη φιλοδοξία. Φανταστείτε ότι η Κομισιόν δεν είχε παρουσιάσει τις προτάσεις που υιοθέτησε στην πλειοψηφία του το Κοινοβούλιο. Τι απάντηση θα μπορούσαμε να δώσουμε στους Βρετανούς φίλους. Θα ήταν ίσως το, το πρόγραμμα της Κομισιόν. Μετά τη Βρετανική ψήφο, θα θέσουμε τέρμα στην προσπάθειά μας. Που όλοι την αναγνωρίζουν, δεν την εκτιμούν όλοι. θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε την γραφειοκρατία στην Ευρώπη. Ήδη προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εμείς στην Κομισιόν είπαμε ότι η κοινωνική Ευρώπη θα βρει μια πραγματική θέση στην Ευρώπη. Ε, τη θέση που της ανήκει. Ξεκίνησα μια ευρεία διαβούλευση για τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα θέλατε η Βρετανική ψήφο να μα φρενάρει, να σταματήσει αυτό. Όχι. Η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει πιο κοινωνική και θα γίνει. Θέσαμε τέλος ω σώμα επιτρόπων σε αυτή την τυφλή μονομέρεια που ήθελε ότι η μόνη απάντηση στην οικονομική και χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση είναι η λιτότητα ελαστικοποίησαμε, αν και δεν τολμώ να πω εύκολα αυτή τη λέξη, ε, το σύμφωνο σταθερότητας. Θέλετε, λόγω της Βρετανικής ψήφου, να επανέλθουμε στην κατάσταση πριν από την ανάληψη των καθηκόντων αυτής της ε, Επιτροπής. Όχι, θα πρέπει το σύμφωνο να εφαρμοστεί με σύνεση και θα το κάνουμε. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για την Ενεργειακή Ένωση. Τι θέλετε, να σταματήσουμε γιατί όλοι λένε όλα. Πρέπει να τα αλλάξατε όλα, χωρί να λένε όμω τι πρέπει να αλλάξουμε, πώ να τα αλλάξουμε. Θέλετε να σταματήσουμε αυτή την συνολική προσπάθεια. Να σταματήσουμε πια να είμαστε εξαρτημένοι από τη Ρωσία. Και να υπάρξει μια ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Όχι, θα συνεχίσουμε προς αυτή την οδό. Θα εξυγχρονίσουμε την Ευρώπη, το είπαμε πολλές φορές. Ακριβώς γι' αυτό ξεκινήσαμε μια φιλόδοξη προσπάθεια για το ψηφιακό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Όχι. Η Κομισιόν θα συνεχίσει προς αυτή την οδό που την ξεκινήσαμε με την αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Όλοι λένε να τα αλλάξετε όλα, αλλά δεν μας λένε τι. Η Κομισιόν όμως αισθάνεται ήρεμη κυρίως χάρη στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αισθάνεται ότι πρέπει να συνεχίσει πάνω σε αυτή την ατραπό που ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο του 2014. Πρέπει όλα να τα αλλάξουμε. Ναι, αλλά όχι το ουσιώδε. Και ποιο είναι αυτό, ότι η Ευρώπη είναι ένα εγχείρημα για την οικοδόμηση του μέλλοντος και της ειρήνης. Αυτό σας το λέω εδώ. Δεν είμαι ούτε κουρασμένος, ούτε άρρωστος, όπως λένε οι εφημερίδες στη Γερμανία. Τώρα οι γιατροί έγιναν και δημοσιογράφοι δηλαδή, ε. Είμαι αυτό που είμαι. Μέχρι την τελευταία μου πνοή θα δώσω μάχη για την Ενωμένη Ευρώπη. Sehr verehrter κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η καιροί είναι πολύ σοβαρή. Ακούω από διάφορες πλευρές ότι θα πρέπει κανείς να αντιδράσει με νυφαλιότητα, να περιμένουμε λιγάκι. Ε, ξέρετε, ε, δεν φαντάζομαι θα εκπλαγεί κανείς από εσά. Εγώ είμαι ψύχρεμο άνθρωπο, αλλά ξέρετε κάτι, εμένα δεν μου αρέσει η ανασφάλεια και θα επιθυμούσα Διακάώ να μας πούν οι Βρετανοί φίλοι μας ε, τι ακριβώς έχουν κατά νου. Την Παρασκευή το πρωί συναντήθηκα με τον πρόεδρο Σούλτς, τον πρόεδρο Τούσκα και τον πρόεδρο Ρούτε και συμφωνήσαμε όλοι μας να παρακαλέσουμε τους Βρετανούς φίλους μας να μας δώσουν αυτό το αίσθημα ασφάλειας το συντομότερο δυνατόν. Και πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει γιατί εγώ ο οποίος από τη Μεγάλη Βρετανία παρουσιάζομαι ως μη δημοκράτης, ως ρομπότ, ως μηχανή, ως γραφειοκράτης, τεχνοκράτης εγώ λαμβάνω υπόψη υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο. Όμω φαίνεται δεν το λαμβάνει η Μεγάλη Βρετανία υπόψη τη. Και αυτό είναι μια εντυπωσιακή αλλαγή κατά τη δική μου κρίση. Ξέρετε, εγώ σέβομαι αυτά που αποφάσισαν οι Βρετανοί και θα επιθυμούσα επίση, γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, και η Μεγάλη Βρετανία να σεβαστεί αυτά που αποφάσισαν οι Βρετανοί πολίτε. και η ε, συνέχεια να ακολουθήσει, να είναι οι αντιδράσει αυτέ που θα έπρεπε να είναι και όχι εδώ να παίζεται αυτό το παιχνίδι Τη της γάτας και του ποντικού. Γιατί αυτό δεν είναι η ερμηνεία της ετοιμιγορίας του λαού. Η ετιμιγορία του λαού ήταν το συντομότερο δυνατόν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα πρέπει να ακολουθήσουν και οι ανάλογες πράξεις. Και θέλω να σας πω και το εξής, και το λέω με απόλυτη σαφήνεια. Εγώ ανθίσταμαι κατηγορηματικά στο γεγονός ότι καταβάλλονται προσπάθειες, ε, ε, πίσω από το ή στο παρασκήνιο, σε σκοτεινά δωμάτια, η Βρετανική κυβέρνηση να ξεκινήσει κάποιες άτυπες διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν θα το επιτρέψω. Και σας λέω, εγώ έχω δώσει μια εντολή εν είδη μουφτή σε όλους τους επιτρόπους ότι δεν θα λάβουν χώρα μυστικές διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν θα συμβεί. Όμως, οφείλουμε βεβαίως να γνωρίζουμε και αυτό το λέει η απλή ε, λογική, ο κοινός νους, ότι με τη Μεγάλη Βρετανία πρέπει να δρομολογήσουμε μια νέα σχέση. Πώς όμως και αμορφή θα λάβει αυτή η νέα σχέση, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τις σκοτεινές προθέσεις των Βρετανών διαπραγματευτών, αλλά από εμάς. Εμείς είμαστε εκείνοι που θα καθορίσουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θέλουμε να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό όνειρο εξακολουθεί να υπάρχει και εμείς πρέπει να εργαστούμε επ' αυτού με επιμονή, με συνέπεια, με ανανεωμένη ενεργητικότητα και δυναμισμό, με αναζωογόνηση των επιθυμιών μας. Δεν είναι η ώρα για ομφαλοσκόπηση ούτε για μας ούτε για τους Βρετανούς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ρίξουμε ένα βλέμμα στο σύνολο της Ευρώπης και αυτό έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά νου. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε πάντα αυτό κατά νου και πάρα θα το πω παρότι πολλοί μου λένε ότι είμαι ένας ξεπερασμένος βεταράνος όμως εγώ θα σας υπενθυμίσω την ημέρα γέννηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα το ξεχάσει κανεί ποτέ αυτό. Ήταν ένα ειρηνικό οικοδόμημα, ένα ειρηνικό εγχείρημα και οι νέοι Βρετανοί, οι οποίοι αποφάσισαν για την παραμονή τη Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προ αυτού απευθυνόμουν, θέλω να σα πω. Ξέρετε, δεν είναι τώρα η στιγμή κατακαιρματισμού τη Υπήρου. Στι αρχέ του 20ου αιώνα είχαμε περίπου ένα 20% Ευρωπαίου στον πλανήτη. Στο τέλο αυτού του πλανήτη, ο αριθμό είναι πολλαπλάσιος. Σίγουρα δεν είμαστε η κυρίαρχη δύναμη, όμως το ποσοστό της Ευρώπης ε, στην παγκόσμια υπεραξία με τις τελευταίες ε, εξελίξεις θα μειωθεί. Είμαστε η μικρότερη ήπειρος του πλανήτη και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Την Ευρώπη δεν πρέπει κανείς να την κοιτάει μόνο αναδρομικά. Αυτά που ίσχυαν για τη γενιά του πατέρα μου δεν ισχύουν πλέον για τους νέους πολίτες. Δεν ισχύουν για αυτούς οι οποίοι αύριο στο μέλλον θα κυβερνήσουν τις χώρες μας. Το μέλλον ανήκει στους νέους της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, το λόγο λοιπόν τώρα έχει εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο ο πρόεδρο τη πολιτική παράταξη, ο κ. Βίμπερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αφήστε με να ξεκινήσω με τα λόγια ενό νέου από τη Βρετανία που είπε ότι ποτέ δεν θα μάθουμε επακριβώ σε ποιο βαθμό θα χάσουμε ευκαιρίε, φιλίε, γάμου και εμπειρίε. Μια ολόκληρη νέα γενιά βρίσκεται σε καθεστώς σοκ. Πάνω από 73% των νέων Βρετανών επιθυμούσαν διακαώς να παραμείνουν στην Ευρώπη. Συνεθλίβησαν οι ελπίδες τους, οι πολιτικοί, αγαπητοί φίλοι, εκείνοι οι οποίοι Εκείνοι λοιπόν οι πολιτικοί που αγωνίστηκαν για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανία είχαν όμως το πλεονέκτημα να ζουν σε μια Ευρώπη χωρίς τύχη, χωρίς εθνικισμού. και είναι εκείνοι οι οποίοι τώρα εγείρουν νέα τύχη. Το δικό μας το μήνυμα σήμερα είναι ότι η νέα γενιά του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να συνεχίσει να μα εμπιστεύεται. Εμεί δεν θα σα εγκαταλείψουμε. Ναι, πράγματι ήταν και είναι η νίκη των λαϊκιστών. Ε, αυτό το έχουμε διαπιστώσει και από τις δύο πλευρές της μάχης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Έχουμε τους δημαγωγούς και από δεξιά και από αριστερά οι οποίοι επιθυμούν να καταστρέψουν την Ευρώπη. Και από την Πέμπτη όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς διακυβεύεται. Το όραμα της συνεργασίας, η, τα τείχη, ο εθνικισμός, η Ευρώπη. Αυτό είναι το διακύβευμα. Και σήμερα ένα πράγμα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Δεν υπάρχει ΕΛΚ, φιλελεύθεροι, πράσινοι, σοσιαλιστές. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Μόνο ένα πράγμα μετράει. Μετράμε εμείς. Εμείς η πλειοψηφία αυτού του κοινοβουλίου τα σώματα υπέρ μιας ενωμένη ειρηνική, ανεκτική Ευρώπης και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι λαϊκιστές. Εμείς στηρίζουμε και θέλουμε αυτή την Ευρώπη σήμερα περισσότερο από ποτέ. και κάποιος άλλος θα πρέπει να μνημονευτεί. Εκείνοι που χρησιμοποιούν κηρύγματα μίσους και χρησιμοποιούν και ψέματα. Το πρώτο ψέμα στο UKIP, στην πολιτική παράταξη UKIP. Την Παρασκευή το βράδυ ο Φάρατς, ο πρόεδρος, είπε ότι είχαν υποσχεθεί 350 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα που τελικά όμως δυστυχώς δεν θα διοχετευτούν στο σύστημα υγείας Μεγάλης Βρετανίας. Ψέμα. Δυστυχώς ψέμα. Κύριε Φάρατς, θα έπρεπε κανονικά σήμερα να ζητήσετε συγνώμη από τους Βρετανούς. Ντροπή σας. Και επίσης ομολογώ ότι και εγώ έκανα ένα λάθος. Και εγώ υπέπεσα στο λάθος να παραμείνω σιωπηλός. Δεν ύψωσα τη φωνή μου, δεν εξέφρασα τη γνώμη μου. Για το μέλλον όμως έχουν περάσει πλέον αυτές οι εποχές εφησυχασμού. Οφείλουμε να στηρίξουμε μαχητικά το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Αγαπητοί λοιπόν συνάδελφοι, σήμερα όταν μιλάμε για μια καλύτερη Ευρώπη, ξέρετε εγώ δεν έχω κατά νου τις μεταρρυθμίσεις, τα τεχνικά. Έχω κατά νου τον David Cameron, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα αγωνίστηκε για την Ευρώπη ως πραγματικός ηγέτης και πολιτικός και αυτό το σέβομαι. Όμως και εκείνος έκανε σταδιοδρομία στην πλάτη της Ευρώπης και των Βρυξελών και άσκησε πίεση στην Ευρώπη. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να εκπλήσεται που οι άνθρωποι δεν τα κατανοούν όλα αυτά. Ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτόν τον τρόπο όμως συμπεριφέρονται πολλοί πολιτικοί από διάφορα κράτη και γι' αυτό σας λέω σταματήστε πια όλοι εσείς αυτό το λαϊκισμό και επιτέλους αναλάβετε τις ευθύνες σας. Η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγές και αυτό δεν το αμφισβητεί κανεί που βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα. Εμεί όμω θέλουμε να βελτιώσουμε και όχι να καταστρέψουμε την Ευρώπη. Γιατί αν καταστραφεί η Ευρώπη δεν θα υπάρχει καμία εναλλακτική λύση παρά μόνο το άσχημο πρόσωπο του εθνικισμού. Οι άνθρωποι λοιπόν στην Ευρώπη πρέπει να γνωρίζουν δεν υπάρχει απόθεμα Ευρώπη, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Το δημοψήφισμα ήταν απόλυτα σαφέ και υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα εδώ Η ε, Μεγάλη Βρετανία δεν έχει ηγεσία, το κόμμα είναι διχασμένο, η, σκοτική, η κυβέρνηση τη Σκοτία εξαιτία ε, διαβουλεύεται για το τι θα γίνει με την ανεξαρτησία τη. Τρία εκατομμύρια Βρετανοί ε, σκέπτονται και επιθυμούν πάλι το δημοψήφισμα, ένα νέο δημοψήφισμα. Δεν υπάρχει λοιπόν σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει το μέλλον. Και μόνο αυτό υποτιμάται η λίρα της Αγγλίας, οι διακοπές για τους Βρετανούς γίνονται πιο ακριβές και αυτό δεν αφορά μόνο τους Βρετανούς. Στην Ολλανδία την Παρασκευή τα συνταξιωτικά ταμεία έχασαν το 3%. Οι Ολλανδοί συνταξιούχοι θα υποστούν περικοπές και αν δεν τους αρέσει παρακαλώ να διαμαρτυρηθούν στον κύριο Φέρετζ. Και στο πλευρό του Φέρετζ βρίσκεται και ο Πούτιν που χαίρεται για όλα αυτά τα αποτελέσματα και αυτά μιλούν όλα από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο. Αγαπητοί λοιπόν συνάδελφοι, η Μεγάλη Βρετανία με αυτό το δημοψήφισμα μόνη της ε, αυτοπυροβολήθηκε. Όλοι οι Ευρωπαίοι βλέπουν πως η Μεγάλη Βρετανία διολυσταίνει σε κρίση, δεν έχει ηγεσία, υφίσταται οικονομικές συνέπειες και ίσως και καταρρεύσει κάτω από αυτό το βάρος. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα του να θέλει κανείς να εγκαταλείψει την Ευρώπη. Όλοι μας οφείλουμε να σεβαστούμε το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπε και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιμένουμε επιτέλους το αίτημα με βάση το άρθρο 50 και να ξεκινήσουν ταχύτατα διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διεξάγει τις διαπραγματεύσεις υπό την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί αν ακολουθήσει μια μακρά περίοδος αυτό θα είναι δηλητήριο. Εμείς χρειαζόμαστε ένα, μια ξεκάθαρη διαδικασία. Ε, όσοι υποστήριξαν την έξοδο υποσχέθηκαν στην Μεγάλη Βρετανία ε, απόλυτη κυριαρχία. Θα αναφέρω εδώ δύο παραδείγματα. Όλοι όσοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους είναι αναγκασμένοι να δέχονται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει για την Ελβετία, ισχύει για την Νορβηγία μα στο μέλλον θα ισχύει και για τη Μεγάλη Βρετανία και το δεύτερο που θέλω να χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα είναι το εξής. Όποιος προσπαθήσει σε Πολωνούς ε, τεχνίτες, ε, σε Ρουμανικές ε, νοσοκόμες, σε Λιτουανούς εργαζόμενους, το μέλλον να τους απαγορέψει την είσοδο στη Μεγάλη Βρετανία, μα αυτός δεν μπορεί να περιμένει στο μέλλον πάλι η Μεγάλη Βρετανία να έχει είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη εδώ δεν έχουμε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, λυπάμαι, αλλά αυτό πρέπει να το κατανοήσει και η Μεγάλη Βρετανία. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ να σας πω σήμερα κατά πόσον το ΕΛΚ θα συμφωνήσει σε αυτό το αίτημα εξόδου. Γιατί ξέρετε, εμείς θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των 44 εκατομμυρίων πολιτών και όχι πια τα συμφέροντα του City του Λονδίνου. Γιατί για μένα, ξέρετε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν επιλέγουμε πια αυτά που μας αρέσουν και αφήνουμε τα άλλα κατά μέρο. Όλες οι κρίσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, εγκυμονούν όμως και ευκαιρίε. Επιτρέψτε μου να επισημάνω το εξή. Από από το 89 οι άνθρωποι στην Ευρώπη διοργάνωσαν 27 δημοψηφίσματα και έδειξαν την προσήλωσή τους στην Ευρώπη. Να καταστήσω σαφές, υπάρχει μια απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών επιθυμούν να βαδίσουν τον κοινό δρόμο προς μια ενωμένη Ευρώπη. Έτσι λοιπόν η απάντηση που θα δώσουμε είναι πάρα πολύ απλή. Οι άνθρωποι περιμένουν από εμάς τους πολιτικούς ταγούς μόνο ένα πράγμα επιτέλους μας λένε κάντε καλά τη δουλειά, τους, δουλειά σας. Σήμερα το απόγευμα θα συναντηθούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και κατά την άποψή μου το Brexit είναι ο συναγερμός για τους αρχηγούς αυτούς γιατί θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε και θα πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι έχουμε ικανότητες ηγετικές. Και αν το κάνουμε αυτό, τότε η Ευρώπη θα στηριχθεί από τους πολίτες της και με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσει στο μέλλον. Και τελειώνοντας, θέλω να επισημάνω εθνικισμός από τη μία Ευρώπη από την άλλη. Πρέπει να σας πω, ξέρετε, η δική μου η πατρίδα είναι η Βαβαρία. Εγώ αγαπώ τη βαβαρική διάλεκτο, αγαπώ την βαβαρική παράδοση και η πατρίδα μου είναι η Γερμανία. Τώρα που παίζει η γερμανική ομάδα στο ευρώ, τρελαίνομαι με την δική μου την εθνική ομάδα. Με την καρδιά και με το νου είμαι πεπισμένος Ευρωπαίος, γιατί αυτή είναι η πυρός μου με μια πολυσχηδή μορφή, μια πολυμορφία στον πολιτισμό και να σας πω κάτι. Κανείς, μα κανένας ακραίος εδώ σε αυτή την Ήπειρο δεν θα μου πάρει τη δική μου την πατρίδα. Εγώ είμαι Βαβαρός, είμαι Γερμανός πολίτης και είμαι ακράδαντα πεπισμένος Ευρωπαίος. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει εκ μέρου ε, των ε, Σοσιαλδημοκρατών ο πρόεδρος της πολιτικής ομάδας, ο κύριος Πιτέλα. Ευχαριστώ, Πολύ σωστά τα είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Κέρδισε τον Brexit. Και πρέπει να δεχτούμε αυτή την ψηφοφορία και το αποτέλεσμά της. Να σεβαστούμε τη θέληση της πλειοψηφίας. Με αυτό το σεβασμό θέλω να σας πω ότι η πρώτη μου σκέψη πηγαίνει σε εκείνους τους Βρετανούς που την Πέμπτη είχαν το κουράγιο και το θάρρος να επιλέξουν την Ευρώπη. Κυρίως στους νέους Βρετανούς που επέλεξαν το μέλλον. Μαζί σας είμαστε. Είμαστε η Ευρώπη του Εράσμους. Είμαστε η Ευρώπη του πολιτισμού. Είμαστε η Ευρώπη η οποία χρηματοδότησε τα καλύτερα ερευνητικά προγράμματα στα Βρετανικά πανεπιστήμια. Είμαστε η Ευρώπη του διαλόγου και του σεβασμού των θρησκειών. Είμαστε η Ευρώπη της ειρήνης. Και η βασική αξία της Ευρώπης είναι αυτή και την έχουν στην καρδιά τους οι νέοι Βρετανοί. Καμία ψήφος, κανένα δημοψήφισμα δεν μπορεί να σπάσει αυτή τη σχέση, αυτόν τον συναισθηματικό δεσμό που δένει το Ηνωμένο Βασίλειο με αυτή την Ήπειρο και λόγω ιστορίας και λόγω πεποίθησης παραμένει τμήμα μιας υπήρου που δεν είναι ή μιας ένωσης που δεν είναι απλώς μια συνθήκη. Και μέχρι να φύγει το ΕΒ οριστικά, αυτός ο οίκος θα είναι οίκος και των Βρετανών. Καταρχάς, οι... αυτοί που πούλησαν φούμαρα, που είπανε ψέμα στους, Βρετανικ... στους Βρετανικούς, είναι υπεύθυνοι και η, απόδειξη είναι μπροστά στα μάτια σα την επόμενη μέρα. Είχαν υποσχεθεί στους εκλογεί διάφορα πράγματα. Οι συντηρητικοί αυτοί οι είχαν υποσχεθεί ότι θα βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πραγματικότητα όμως αφήσανε ερήπια. Μια φοβερή συνταγματική κρίση με τη Σκοτία. Ένα πολιτικό χάος σε όλη τη χώρα την κατάρρευση της Τερλίνας. Μια πραγματική ε, ζημιά στην πραγματική οικονομία. Και αφού κατέστρεψαν τη χώρα, κάποιοι θέλουν τώρα να καταστρέψουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να παραλύσουν την θεσμική τη ζωή. Εγώ θέλω να σας πω ξεκάθαρα, δεν μπορεί να γίνεται όμπειρος των ε, παιχνιδιών, των εσωκομματικών παιχνιδιών των Βρετανών, των κομματικών τεχνιδιών των Βρετανών. Και οι ευρωπαϊκές και φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις που κατοικούν και δρεύουν εδώ θα αντιμετωπίσουν με αραγές μέτωπο όλη αυτή την προσπάθεια. Για να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε και να σώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αγγλικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν τη θέλησή του για να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις αμέσως μετά την κοινοποίηση αυτή. Εγώ θα ήθελα να σας καλέσω να κάνουμε ένα πιο βαθύ προβληματισμό, αγαπητοί συνάδελφοι. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν είναι μόνο αποτέλεσμα μιας ρώσικης ρουλέτας, της ρώσικης ρουλέτας που έπαιξε ο Κάμερον. Η παγκοσμιοποίηση δημιούργησε μιας καταστάσει, κάποιες καταστάσεις, κάποιους νικητές και κάποιου ηττημένου. Κάποιε ανισότητες. Και εμείς ήμασταν πολύ δειλοί να υπερασπιστούμε του ηττημένου και να του διασώσουμε. Πιστεύαμε ότι η αγορά θα μπορούσε να τα σώσει, να σώσει τα πάντα. Ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει τρομερά πράγματα. Εγκαταλείψαμε τους εργαζόμενους. Ε, εγκαταλείψαμε την ιδέα της ισότητας. Οι χρηματαγορές είχαν την απόλυτη εξουσία, οι οποίοι τελικά έκαναν κακό και στη δημοκρατία και στην πολιτική και στα θεσμικά όργανα. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο κάναμε τη δουλειά μας. Κάναμε μια προσπάθεια για την Τραπεζική Ένωση, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για να διατρανώσουμε τη δύναμη της ε, δημοκρατίας πάνω σε αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις των ε, χρηματοπιστωτικών κύκλων που σκοτεινά δουλεύουν. Έχουμε μία Ήπειρο διαιρεμένη. Έχουμε μίσος, έχουμε απελπισία στην Ήπειρό μας. Και μπορεί να παρασύρει τα πάντα. Η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν. Και η πρώτη ερώτηση και η πρώτη απάντηση την είπε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Σεβασμό στη δικαιοσύνη. Και όταν μιλάω για δικαιοσύνη, μιλάω για άτομα, μιλάω για ανθρώπους. Δικαιοσύνη κοινωνική. Αναθεώρηση της οδηγίας απόσπασης των οδηγών, ε, των εργαζομένων. Καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ή θα συνεχίσουμε έτσι, ή θα αφήσουμε ανοιχτό το δρόμο για να πολεμήσουμε μεταξύ τους οι φτωχοί. Επίσης, υπενθύμισε διάφορα πράγματα ο Γιούνκερ για το δημοσιονομικό σύμφωνο. Εμεί ω σοσιαλιστέ θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να υπάρξουν δημόσιε επενδύσει. Ιδιωτικέ επενδύσει επίση φυσικά. Πρέπει να υπάρξει ένα πιο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο. Και το λέω σήμερα ότι η ομάδα μα θα αντιταχθεί στην, στο να υπάρξει μόνο το δημοσιονομικό σύμφωνο και μέχρι εκεί να σταματήσουμε. Θα πρέπει να το μετασχηματίσουμε, να το αλλάξουμε άρδιν. Εγώ δεν το υπερψήφισα. Δεν το υπερψήφισα το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Πηγαίνετε να διαβάσετε πριν μιλάτε έτσι. Να καταπολεμήσουμε αμήλικτα τους φορολογικούς παραδείσους, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Να εφαρμόσουμε τα μέτρα που ενέκρινε η Επιτροπή Τάξε Υπάρχει το μεγάλο θέμα επίση τη δημοκρατία. Κάθε πολίτη θα πρέπει να μετράει. Εμεί προτείνουμε στι επόμενε ευρωπαϊκέ εκλογέ να προβλέψουμε άμεση εκλογή του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αρχηγό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Δήμαρχο Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να έχουν μπροστά του το ψηφοδέλτιο το όνομα αυτού του ανθρώπου που θα είναι ο αρχηγός. Αυτό σημαίνει να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό πολιτικό χώρο ευρωπαϊκής φύσεως. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρο να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς εκλεγήκαμε απευθείας από του πολίτες που πιστεύουν στην Ευρώπη και θα πρέπει να πολεμήσουμε κάθε δύναμη με το συνέστημά μας, με το πάθος μας, για να μην προδώσουμε τους πολίτες που μας διάλεξαν και μας υποστήριξαν. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καμάλ τώρα, επικεφαλής της ομάδας ECR. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Οι Βρετανοί μίλησαν και ψήφισαν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιες και αν είναι οι δικές μας προσωπικές πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση αυτή του Βρετανικού λαού και να προχωρήσουμε μπροστά. Φυσικά, πολύ συναισθηματισμός και από τις δύο πλευρές της μάχης. Υπήρξε η προεκλογική εκστρατεία και πολλοί έχουν πει ότι η Βρετανή πολιτική θα έπρεπε να είναι πιο ειλικρινής όσον αφορά την πολιτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Άνωσης. Και τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις με, τον, με τους Βρετανούς. Αυτά είναι στο παρελθόν. Τώρα πια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να στραφούν προς το μέλλον. Και από τις δυο πλευρές πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε την διαπραγματευτική μα στρατηγική. έχει πρόθεσμα να δούμε πώς μπορούν να υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, το είπε και η Ολλανδική Προεδρία. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιε θα είναι οι σχέσει αυτέ με το Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλοι λένε να πάμε αργά. Άλλοι λένε να τιμωρήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλοι λένε μα ε, εμεί θα αποφασίσουμε. Οι διαφορέ που υπάρχουν υπάρχουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά πόσο θα ενεργοποιηθεί γρήγορα το άρθρο 50. Αν τη συμφωνία θα υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια μορφή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ξεκάθαρη, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο από τη δικιά του την πλευρά επίση. Συγχρόνω. Όμως η απόφαση είναι απόφαση και πρέπει να γίνει σεβαστή. Οι διαπραγματευτές από όλε τις πλευρές πρέπει να προσφέρουν βεβαιότητα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να προετοιμαστούμε έτσι ώστε όταν αναργοποιηθεί το άρθρο 50 να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και πρέπει αυτές να είναι υποφελείς και για τις δύο πλευρές. Αυτό που έχει συμφωνία είναι η τελική συμφωνία στην οποία θα καταλήξουμε και όχι το πότε θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Για αιώνες υποδεχόταν το Ηνωμένο Βασίλειο ανθρώπους από ολόκληρο το κόσμο και όταν υπήρχε φασισμός ε, αλλού ανοίξαμε τις πόρτες μας. Υποδεχτήκαμε όλους τους λαούς και όλα έθνη και θα παραμείνουμε ένα ανοιχτό έθνος. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να είναι εταίροι και τις επόμενες δεκαετίες. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Συνεπώς τώρα μην κοιτάμε πια στο παρελθόν, ας κοιτάμε προς το μέλλον. Ας φροντίσουμε να σκεφτούμε τις διαπραγματεύσεις και εμείς οι Βρετανοί θα είμαστε καλοί γείτονε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εκ μέρους των φιλελεύθερων, ο πρόεδρος Φεχόστατ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω στρεφόμενος προς τους Βρετανούς και να τους πω ότι είναι πάντα σκληρό να δέχεται κανείς μια απόφαση με την οποία διαφωνεί. Αλλά πρέπει να τη δεχτούμε. Η επιλογή ήταν σαφής. Πρέπει να τη σεβαστούμε. Τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούν τουλάχιστον 700 ευρωβουλευτές εδώ. Το θέμα δεν είναι τόσο η επιλογή που είναι σκληρή. Είναι μια επιλογή. Μια επιλογή, εντάξει, αυτή είναι και η ουσία της δημοκρατίας, κάθε δημοκρατίας. Αυτό όμω που είναι τόσο δύσκολο για μένα, τόσο σκληρό, αλλά και για τους άλλους επικεφαλής ομάδων εδώ, αλλά και για τους υπόλοιπου, είναι ο τρόπος με τον οποίο φτάσαμε σε αυτή την απόφαση. Μια πολύ αρνητική προεκλογική εκστρατεία. Τα πόστερ, ε, οι αφήσει του κύριου Φαράτζα δείχνανε μετανάστες συνδεδεμένους με την ε, ναζιστική προπαγάνδα. Δεν ήξερα ότι θα μπορούσε κάποιος από αυτό εδώ το σώμα να κάνει κάτι τέτοιο. Τα ψέματα για τη μετανάστευση τα ψέματα για την Τουρκία που θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεθαύριο. Ή τα ψέματα για τα 350 εκατομμύρια λίρες που αμέσως θα επέστρεφαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και τώρα, α, δεν γίνεται. Αυτό το κλίμα φόβου, αρνητισμού που δημιουργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι που με σοκαρεί περισσότερο για το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι επιλογή του κόσμου, γιατί η επιλογή του κόσμου είναι η δημοκρατία. Και σήμερα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Βλέπουμε να χάνονται δισεκατομμύρια στις ε, αγορές, στο χρηματιστήριο, πέφτει η λίρα. Τώρα που θα μιλήσετε, περιμένετε, θα δείτε, θα κατέβει κι άλλο μόλις πάρετε το λόγο η λύρα, κύριε Φάρατς. Και κάθε φορά που μιλάει ο Μπόρις Τζόνσον χειροτερεύει η κατάσταση. Οπότε το Brexit, να το. Ο κύριος Καμάλ λέει, «Ε, όχι προσωρινά, έτσι για λίγο. Δεν ξέρω. Μακάρι. Αλλά αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι όσο γίνεται πιο γρήγορα πρέπει να σταματήσει αυτή η περίοδος αβεβαιότητας. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε τώρα. Και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να συνεχιστεί η αβεβαιότητα. Μόνο η ιδέα για την αποχώρηση μπορεί να σταματήσει αυτό το κλίμα αυτό το τοξικό κλίμα το οποίο δημιουργείται. Όμως, κύριε Φάραντς, η δουλειά που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει για τους αξιοπρεπείς, κύριε Φάραντς. Η ενεργοποίηση λοιπόν του περίφημου άρθρου 50 δεν είναι τιμωρία. Κάθε άλλο θα έλεγα εγώ. Σημαίνει ότι σεβόμαστε την επιλογή του κόσμου η ενεργοποίησή του, αλλά είναι μια πράξη που δεν θέλει η ηγεσία των τόρις. Ένας είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα, ακόμα και να θυσιάσει τη φωνή 700 εκατομμυρίων, 70 ε, εκατομμυρίων Βρετανών. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμείς, λοιπόν, και το λέω αυτό σε όλους τους συναδέρφους, ότι οι Βρετανοί Ευρωπαίοι δεν μπορεί να θυσιαστούν και να βρεθούν σε αυτή την αβεβαιότητα. Ο κ. Καμαλιά πρέπει να διαπραγματευτούμε, να προετοιμαστούμε κτλ. Πώς είπατε, να προετοιμαστούμε, μα κέρδισε το Λιβ, κύριε Καμάλ. Ο κύριος Καμάλ λέει δεν ψήφισε για το Λιβ. Οι άλλοι, Βρετανοί. Συνεπώς, εμείς, οι 27 υπόλοιποι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να περιμένουμε για ένα κόμμα των τόρις από προσανατολισμένο μέχρι να συνέλθει. Όχι. Πρέπει να προχωρήσουμε με θάρρος, με πεποίθηση, ενωμένοι προς ένα νέο ορίζοντα. Γιατί υπάρχει νέο ορίζοντα, υπάρχει νέο μέλλον για την Γυρέπηρο και για να τα καταφέρουμε Πρόεδρε, θα σας πω και θα το πω σε όλου του συναδέρφους ότι δεν χρειαζόμαστε και πολύ φαντασία. Ξέρετε τι χρειαζόμαστε. Να θυμόμαστε. Μνήμη χρειαζόμαστε. Καλή μνήμη για να επανέλθουμε στις αρχικές ιδέες των ιδρυτών πατέρων. Αυτό χρειαζόμαστε. Και σήμερα είναι ξεκάθαρο το τι σημαίνει αυτό jean Κλοντ, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή κυβέρνηση για την Ευρωζώνη. Χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή ακριβώς για να φροντίζει να μπορεί η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών μας να είναι πραγματικότητα. Πρέπει να είμαστε σε θέση να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία και να έχουμε μια κοινότητα Άμυνα όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί οι Αμερικανοί δεν είναι πια ε, διατεθειμένοι να πληρώνουν. Ένα πράγμα χρειαζόμαστε λοιπόν. Όχι να αρχίσουμε επίσημες διαπραγματεύσεις, να προετοιμαστούμε κτλ. Όχι, πρέπει να δείξουμε στους λαούς της Ευρώπης ότι είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ένωση η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει τις διάφορες κρίσεις. Με δύο λόγια, και θα ολοκληρώσω με αυτό. Ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε. Κατ' εξαίρεση, να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή, την εξουσία του σώματος αυτού που είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, προκειμένου να βάλουμε και πάλι την Ευρώπη πάνω στις ράγες. Αυτό και μόνο πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Für die Fraktion der Vereinigten Εκ μέρους της ε, Ενωμένης Αριστεράς η πρόεδρος κυρία Τσίμα. Κοιτάξτε, εγώ τάσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ των δημοψηφισμάτων, όμως τα δημοψηφίσματα πρέπει να οργανώνονται υπεύθυνα και ανάλογη να είναι και η στάση μετά το, την έκβασή τους. Για μένα τα δημοψηφίσματα είναι σαφώς ένα δημοκρατικό εργαλείο. Κατόπιν τούτου το Βρετανικό δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία δεν ήταν απλά η έκφραση βούλησης του Βρετανικού λαού. Πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Όμως είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η Βρετανία αποφάσισε αποφάσισαν και ας κάνουν τώρα ό,τι νομίζουν. Δηλαδή ε, να πιστεύουμε απλά ότι ο σειρμός, ε, το καραβάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσει να μετακινείται. Τα πλασίμπο τα υποκατάστατα φαρμάκων δεν βοηθούν όταν είναι άρρωστος ο ασθενής. Όταν λοιπόν ε, πρόκειται για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας ε, πολλοί επιθυμούν να υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών και γι' αυτό το λόγο όμως εμείς ε, δεν συμφωνούμε δεν συμφωνούμε με το ψήφισμα γιατί θεωρούμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει αυτοκριτική. Κανείς δεν μοιάζει να περισυλλογίζεται και όταν μιλάει κανείς για μνήμες θα πρέπει να έχει κατά νου και άλλες ιστορικές μνήμες, δηλαδή τις λανθασμένες εξελίξεις, ε, τις λάθος υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δεκαετίες. Και δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά τα ίχνη, βαθιά ίχνη που έχουν απομείνει μετά από όλους αυτούς τους ε, χειρισμούς με την Ελλάδα, με την Ιταλία, με όλες αυτές τις χώρες. Μα τι άφησαν όλα αυτά στον Ευρωπαίο πολίτη. Οι συνέπειες της βαθιάς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι συνέπειες αυτές εγχαράχθηκαν στη συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη. Εθνικά κοινοβούλια, κυβερνήσεις, ε, ακόμα και συντάγματα, όλα αυτά αγνοήθηκαν και αυτό ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο. Και δυστυχώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι υποστηρικτές του Brexit ε, είναι εκείνοι οι οποίοι επίσης ανησυχούν για τη θέση τους και για πάρα πολλά άλλα ε, συμπαρομαρτούντα για το συνταξιδοτικό, για το ασφαλιστικό. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα ότι θέλει να προστατεύσει τους ανθρώπους από τις επιπτώσεις της παγκοσμίας παγκοσμιοποίησης. Και ρωτώ, μα πόσο ε, πολύ εθελοτυφλούν τα μέλη του Συμβουλίου που ήδη παλαιότερα είχε ανακοινώσει ο Κάμερον ότι επιτιμούσε να περικόψει τα επιδόματα για τους αλλονταπούς πολίτες και πώς μπορούν να μην γνωρίζουν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτό θα αφορούσε πάρα πολλούς Βρετανούς πολίτες και οι θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ συμπεριλαμβάνω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι θεσμοί λοιπόν επέτρεψαν η θέση τη Μάργαρετ Θάτσερ που ήταν ότι ξέρετε δεν υπάρχει κοινωνία είχε πει η Θάτσερ αυτή η πολιτική μοιάζει να επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αλληλεγγύη, οι κοινοτικέ μέθοδοι αυτά έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Άγγελα Μέρκελ και είναι εξίσου όπως και άλλες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, παραδείγματος χάρη η κρίση του προσφυγικού και όλες οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση σε συνδυασμό με τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτά λοιπόν προκάλεσαν φόβους, φόβοι οι οποίοι στράφηκαν κυρίως ε, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα πράγμα θέλω να σας πω. Αν ως Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αντίδραση της Βρετανικής ελίτ και είχαμε ζητήσει ίδιο μισθό για ίδια εργασία, αν τα είχαμε κάνει όλα αυτά, τότε δεν θα είχε υπάρξει αυτή η διασύνδεση ανάμεσα σε φόβους μισθού και θέσεων εργασίας και πρόσφυγες. Κύριε Φαράτζ, ανεξάρτητα με το τι εντύπωση θέλετε εσείς να προκαλέσετε, θέλω να σας πω ότι με την εκστρατεία σας ε, ποτέ δεν μπορέσετε να ξεπεράσετε το μικρό το φοβικό. Και το πρόβλημα είναι ότι ένα κομμάτι της πολιτικής και οικονομικής ελίτ του Λονδίνου αντέδρασε, διαφώνησε και θέλησε να πείσει ότι εσείς επιθυμείτε μια νέα νεοφιλελεύθερη τάξη στην Ευρώπη. Και ξέρετε, η ιστορία θα διατηρήσει το όνομά σας, θα παραμείνετε με αυτή την εικόνα στην ιστορία, όμως εγώ οφείλω να επισημάνω ότι αυτά που είπατε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας σας ε, για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες, απλά υποδάβλησαν το μίσος. Ε, εγώ δεν θέλω να ε, επικρατεί άποψη ότι θέλουμε να τιμωρήσουμε τους Βρετανούς. Όμως πρέπει να υπάρχει και σαφήνεια. Δεν μπορεί να υπάρχει σαφήνεια όσο η ε, Μεγάλη Βρετανία δεν έχει επικυρώσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Εξάλλου, εμείς θεωρούμε ότι η πλειοψηφική απόφαση των πολιτών στη Σκοτία και στην Βορειολανδία και αυτή θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Δεν θέλουμε να απαλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ευθύνες της. Ε, επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναλάβει μόνη της την επίλυση του θέματος ε, της Βόρειας Ιρλανδίας. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη στους πολίτες επιτόπους. Σήμερα λοιπόν τίθεται το θέμα της διαδικασίας. Εμείς ε, επιθυμούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή εξ αρχής ε, να συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις και όχι μόνο όταν θα έχει ληφθεί η απόφαση για τη συνθήκη και επιθυμούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει ευθύ εξ αρχής όταν θα τεθούν τα περαιτέρω θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν διαπραγματεύσεις να γίνονται και κλεισμένων των θυρών και το πρώτο βήμα που πρέπει να λάβει η χώρα είναι επιτέλους να συμβάλλετε και εσείς έτσι ώστε αυτή η ολέτρια κοινοτική μέθοδος να αντικατασταθεί επιτέλους από την διακυβερνητική μέθοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των ε, Πρασίνων, ε, ο κύριος Λάμπερτς. Συνάδελφοι, υπάρχουν κάποιες στιγμές όπου η πολιτική ο πολιτικός χρόνος εωρείται και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια επιλογή. Την ε, επαύριο του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, τα κράτη είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν ή να σπάσουν την αρχή της εθνικής κυριαρχίας. Αποφάσισαν να επιμεριστούν αυτή την ε, κυριαρχία και γι' αυτό εξασφάλισαν μία ε, περίοδο ειρήνης και ευημερίας χωρίς προηγούμενο στην ε, ευρωπαϊκή ιστορία. Η απόφαση του δημοψηφίσματος της, ε, του Μεγάλου Βασιλείου σπάει αυτή την ε, συνέχεια. Η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Γαλλία κτλ. Σε όλες αυτές τις χώρες βλέπουμε σημάδια ανησυχίας των λαών στην, και αμφισβήτησης της ευρωπαϊκής αυτής διαδικασίας. Και ακόμα τώρα Υπάρχει μπροστά μα, ορθώνεται μπροστά μα μία επιλογή. Και από αυτήν εξαρτάται η επιλογή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τρει επιλογέ. Πρώτον, αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να επανέλθουμε στους εθνικισμούς, ε, στους εθνικισμούς που λέει ο Ορμπάν, ο Φάρατζ, η Λεπέν κτλ. Όλοι αυτοί. Και να, σου... να κλειστούμε πάλι στον εαυτό μας. Στου... Τους λέω το εξής. Έχετε δίκιο. Πρόκειται για την ε, δημοκρατική κυριαρχία, για την ικανότητα των δημοκρατιών μας να κάνουν ελεύθερα επιλογές για να καθορίσουν το μέλλον τους. Αλλά λέτε και ψέματα. Λέτε ψέματα. Γιατί ποιος μπορεί να πιστέψει ότι το πιο ισχυρό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί από μόνο του και επιτυχώς να ανταπεξέλθει στη φοβερή ε, απειλή των ε, πολυεθνικών, στο οργανωμένο έγκλημα, στην αλλαγή του κλίματος στο μεταναστευτικό, στο προσφυγικό. Κανένα τείχο δεν θα είναι αρκετά ψηλό ή αρκετά παχή για, για να απομονώσει την Ευρώπη από τι προκλήσει του 21ου αιώνα. Μόνο χάρη στην επιμερισμένη αυτή εθνική κυριαρχία. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε, κύριε Γιούνκερ, είναι αυτή που υπερασπίζονται σήμερα οι περισσότερε ευρωπαϊκέ κυβερνήσει και που υπερασπίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, να εξασφαλίσουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να έχουμε δημοσιονομικούς κανόνες και λογιστικούς κανόνες, ε, οικονομικά λογικούς. Εσείς λέτε να επαλευθερώσουμε τις α, δυνάμεις της αγοράς, να επιμένουμε με αρρώστια, κυρία Μάτσομ, να φτιάχνουμε εμπορικέ συνθήκε, υποτίθεται, όπου ο βασικό στόχο είναι στην πραγματικότητα να λησοδέσουν τι δημοκρατίε μα. Συχνά προ προτιμούμε την αδιαφάνεια, και εδώ στρέφουμε προς το Συμβούλιο, από την διαφάνεια στις αποφάσεις. Προκειμένου να πληρώσει το πολιτικό τίμημα των αποφάσεων. Αυτή την πολιτική επιβάλλουμε στην Ευρώπη εδώ και 25 χρόνια. Γιατί κύριε Γιούνκερ τότε επιλέξατε, μια και θέλετε συνέχεια, δεν είχατε πει ότι θα ήσασταν πρόεδρος της Κομισιόν. όσοι θέλουν αυστηρή νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία τους λέω ότι το να αλυσοδέσετε τα κράτη-μέλη δεν δίνει ανάπτυξη. Ανάπτυξη δεν δίνει μείωση των ανισοτήτων και το να κάνουμε τους πλούσιους πιο πλούσιους δεν προωθούν την ισότητα. Ακριβώς γι' αυτό αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός, γιατί αφήνει στο περιθώριο όλο και περισσότερους συμπολίτε μας. Εμείς, εμείς θέλουμε να επιλέξουμε μια τρίτη οδό και φιλοευρωπαϊκή, καμία αφιβολία γι' αυτό, θέλουμε να σπάσουμε αυτή την ενιαία και ορθόδοξη σκέψη. Θέλουμε να επανέλθουμε στι ρίζε του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, που ήταν να εξασφαλίσουμε την ε, ειρήνη, να υπάρξει μια φιλελεύθερη ελευθερία ε, ακόμα πιο μεγάλη και, μια, ε, και ένας πλούτος και μια ευημερία που να, την, να είναι ανοιχτή για όλους. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του Ευρώπη μέσω μιας πραγματικής δημοσιονομικής ένεσης θα μπορούσαμε να κάνουμε την ε, Ενεργειακή Ένωση ε, βασικό μας στόχο. Μπορούμε να απαγορεύσουμε τα ψάρια τα οποία τα δηλητήρια τα οποία ε, σπάνε και διαλύουν το περιβάλλον μας. Μπορεί η Ευρώπη να ξαναγίνει χώρα υποδοχής για όλους όσους φεύγουν από τη φτώχεια, τον πόλεμο και τη δίωξη. Μπορούν οι κοινωνίες μας να ζήσουν μέσα στα όρια του πλανήτη μας. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη δημοκρατία μας με μεγαλύτερη διαφάνεια. Με δύο λόγια. Μπορούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων, όλων, και των σημερινών γενιών και των επόμενων γενιών στο κέντρο της πολιτικής. Εμείς λέμε ναι, όλα αυτά γίνεται να τα κάνουμε. Φτάνει να το θέλουμε. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράσει αυτή την πολιτική βούληση τότε θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Εάν αγνοήσουμε τα σημάδια του Βρετανικού δημοψηφίσματος, θα καταστραφεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη έχει γνωρίσει φοβερές τραγωδίες. Πρέπει λοιπόν να ελπίζει, αλλά και να προσπαθεί να οικοδομήσει το καλύτερο. E Εκ μέρου ε, τη ε, πολιτική ομάδα EFDD, το λόγο έχει ο κύριο Φάρατζ. Καλημέρα. Καλή σα ημέρα. Πλάκα έχει. Δεν έχει πλάκα. Όλο αυτό δεν έχει πλάκα. Πρόεδρος, Κύριε Φαράτζ, διακόπτει ο πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, μία, ένα χαρακτηριστικό της δημοκρατίας, καθοριστικό, είναι ότι ακούει κανείς και εκείνους με τους οποίους διαφωνεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σουλτ. Κοιτάξτε, έχει πλάκα γιατί όταν ήρθα εδώ πριν από 17 χρόνια και είπα ότι ξέρετε θέλω να ηγηθώ τη εκστρατεία για να εγκαταλείψει η Μεγάλη Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε όλοι Γελάσατε. Τώρα όμως δεν βλέπω να γελάτε, έτσι δεν είναι. Και ο λόγος που είναι, που είσαστε τόσο αναστατωμένοι και οργισμένοι είναι απόλυτα σαφής. Από όλα αυτά τα οργισμένα που άκουσα σήμερα, ότι εσείς ως πολιτικό εγχείρημα αμφισβητήστε. Αμφισβητήστε εσείς, αμφισβητείτε το νόμισμά σας. Κοιτάξτε, για δέστε λιγάκι τη Μεσόγειο. η πολιτική που επιβλήθηκε για να επικρατήσει φτώχεια στην Ελλάδα και τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Αλλά αμφισβητήστε και με την έκκληση της κυρίας Μέλκεν πέρυσι να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τη Μεσόγειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό οδήγησε σε μεγάλη ένταση ανάμεσα στις χώρες. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε και ο κύριος από χρόν λόγος γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε ως ψήφισε είναι ότι εσείς με απάτες, ε, με ε, ψέματα. Ποτέ δεν είπατε την αλήθεια στους Βρετανούς και στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Τους επιβάλλατε πολιτική ένωση τους επιβάλλατε πολιτική ένωση και όταν οι πολίτες το 2005 στην Ολλανδία και στη Γαλλία καταψήφισαν αυτή την πολιτική ένωση όταν απέρριψαν το Σύνταγμα εσείς απλά ε, τους αγνοήσατε και τι κάνατε από την πίσω πόρτα φέρατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό που έγινε την Πέμπτη ήταν αξιοσημείωτο, ήταν σεισμικό το αποτέλεσμα. Δεν ήταν μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί αυτό που έκαναν οι απλοί άνθρωποι, ο απλό κανονικό μέσο άνθρωπο, ο οποίο τα τελευταία χρόνια πιέζεται και βλέπει να επιδεινώνεται το βιωτικό του επίπεδο, ο άνθρωπο αυτό απέρριψε τι πολυεθνικές, τι συγχωνεύσει τραπεζών, τι μεγάλε πολιτικέ, και είπε αυτό ο απλό άνθρωπο, ξέρετε κάτι, εμεί θέλουμε πίσω πίσω την πατρίδα μας. Θέλουμε πίσω τη δική μας την αλία, τα δικά μας τα σύνορα. Θέλουμε να είμαστε μια ανεξάρτητη, αυτοδιαχειριζόμενη, αυτοδιοικούμενη χώρα. Και αυτό λοιπόν πρέπει να λάβει χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει. Και με τον τρόπο αυτό πλέον δώσαμε αχτίδα ελπίδας ε, στους δημοκράτες και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα κάνω μία πρόβλεψη. Ξέρετε, η Μεγάλη Βρετανία δεν θα είναι το τελευταίο κράτος το οποίο θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή τίθεται το εξή ερώτημα. Και τι θα ακολουθήσει τώρα εναπόκειται στην ε, Βρετανική κυβέρνηση να ενεργοποιήσει το άρθρο 50. Και εγώ θέλω να σας πω ότι εντάξει δεν πρέπει να καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Συμφωνώ με τον κύριο Γιούγκερ ότι εν πάση περιπτώσει η Βρετανία αποφάσισαν τώρα να ακολουθήσουν οι πράξεις. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια όρημη, ευαίσθητη στάση απέναντι σε μια διαφοροποιημένη σχέση. Γνωρίζω ότι κανείς από εσάς ε, στη ζωή σας δεν έχετε κάνει ποτέ μια κάποια δουλειά. Δεν έχετε δουλέψει ποτέ για κάτι σωστά. Ή έχετε, είτε έχετε εργαστεί στις επιχειρήσεις, είτε έχετε εργαστεί στο εμπόριο, είτε έχετε δημιουργήσει μια θέση απασχόλησης. Ποτέ δεν έχετε λειτουργήσει σωστά. Όμως, ακούστε με, πρόεδρος Διακόπτη, κύριε Φάραντζ, αγαπητοί συνάδελφοι, με κάθε σεβασμό για την αναστάτωσή σας. Ξέρετε, εδώ συμπεριφέρεστε σήμερα όπως κανονικά συμφέρεται το κόμμα του κύριου Φάρατζ, το UKIP. Άρα δηλαδή μην μιμήστε τον κύριο Φάρατζ και το κόμμα του. Κύριε Φάρατζ, θέλω όμω να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι εδώ σε αυτή την αίθουσα ε, δεν έχουν κάνει ποτέ μία κανονική δουλειά. Κοιτάξτε, μην κρίνετε εξιδίων τα αλότρια. Δεν ισχύει. Έχετε απόλυτα δίκιο κύριε Σούλτ, ε, λέει ο κύριο Φάρατζε. Εσεί ε, περασπίζασταν ε, το κατεστημένο και τώρα όμω αντιδρά το κατεστημένο. Λοιπόν, α δούμε την πραγματικότητα και τα οικονομικά στοιχεία. Κοιτάξτε, ανάμεσα στι δικέ σα τι χώρε και στη δική μου τη χώρα υπάρχουν πάρα πολλέ ανταλλαγέ εμπόρων, ευμάτων και υπηρεσιών. Αυτό το εμπόριο είναι υποφελέ και για τι δύο πλευρέ και παίζει ρόλο. Εάν λοιπόν πρόκειτο να αποφασίσουμε αποφασίσετε να απορρίψετε οποιαδήποτε ιδέα λογικών εμπορικών ανταλλαγών, τότε οι συνέπειες θα ήταν πολύ χειρότερες για εσάς από ό,τι για μας. Θα ήταν σαν να φτύνατε μόνοι σας το πρόσωπό σας. Και καμία συμφωνία αν θέλετε αυτό είναι πολύ καλύτερο για την Ευρωπαϊκή, για τη Μεγάλη Βρετανία με συγχωρείτε, για τη Μεγάλη Βρετανία από τις συμφωνίες που υπάρχουν τώρα γιατί υπάρχουν συμφωνίες όπου αν ε, εφαρμοστούν, αν δηλαδή επιβληθούν δασμοί, τότε πολλές χιλιάδες Γερμανοί εργαζόμενοι θα χάσουν την εργασία τους στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε ρεαλιστές, ας είμαστε πραγματιστές και ας αποφασίσουμε για μια συμφωνία λογική, χωρίς δασμούς και μετά, μετά τότε πράγματι να αναγνωρίσετε κι εσείς ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι φίλο σας, θα έχει εμπορικές ανταλλαγές με εσά, τότε θα είμαστε ο καλύτερό σας φίλο στον κόσμο. Όμως να γίνουν όλα αυτά λογικά και να μας ε, επιτρέψετε να προχωρήσουμε εμείς και να καθορίσουμε μόνοι μας τα οράματά μας, τις φιλοδοξίες μας και το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το, την πολιτική παράταξη ΕΝΕΦ, e το λόγο έχει η πρόεδρος κυρία Λεπέν. Και όμως, και όμως αγαπητοί συνάδελφοι, μα γιατί εκνευρίζεστε. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι η ιστορία όταν η ελευθερία υπερέχει και θριαμβεύει η βούληση ενός λαού. Η ψηφοφορία των Βρετανών για να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ενωμένο Βασίλειο είναι το πιο σημαντικό πολιτικό γεγονός που έλαβε χώρα στην Ήπειρό μας μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Και είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά είναι και μια κραυγή αγάπης των Βρετανών για τη χώρα τους. Επέλεξαν αυτό που επέλεξαν, μια και να αφήσουν απ' έξω, είσαστε κι εσείς μέσα σε αυτούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδειξαν κατάφορα με αυτήν την τεράστια νίκη τους ότι θέλουν τη δημοκρατία. Είναι ένα χαστούκι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στο φόβο, στον εκβιασμό και στο ψέμα. Στην κραυγή και δώσατε ένα παράδειγμα πριν από λίγο και εσείς ήδη στις απειλές για αποκάλυψη. Πέφτουν τα χρηματιστήρια. Μα οι Βρετανοί αδιαφόρησαν για αυτά και παραμένουν κυρίαρχοι. Κερδίζουν και πάλι την κυριαρχία τους παρά τη δικιά σας έκπληξη. Στο κάτω-κάτω τι είναι αυτό που σας εκπλήσει εσάς. Εδώ και δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικοδομηθεί σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Όντω το γαλλικό και το ολλανδικό δημοψήφισμα τι έδειξαν. Δεν ήθελαν. Παρόλα αυτά μετά αναγκάστηκαν και στο άλλο δημοψήφισμα που έκανε η Ελλάδα οι Έλληνες επειδή τους εκβίασαν να αρνηθούν το αποτέλεσμα του δικού τους του δημοψηφίσματος. Και τώρα έσπασε από τους Βρετανούς η αλυσίδα που τους ένωνε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και που είχε ε, ανεγερθεί σε θρησκεία. Άλλαξαν όλα αυτά που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες με ανόητες παράλογες πολιτικές που οδήγησαν σε μαζική ανεργία, μαζική μετανάστευση. Ε, βέβαια, πόσο δύσκολο είναι κανείς να δει την πραγματικότητα και να αντιληφθεί τι συμβαίνει σήμερα. Όλοι αυτοί οι προπαγανδιστές από την Ευρωπαϊκή Ένωση αριστερή υποτίθεται ή του κέντρου ή της δεξιάς. Ε, λοιπόν τώρα, να, στα μούτρα σας. Τι θα κάνετε, την οργή σας. Δώστε την, κάντε την πάντα και χαρείτε για την απόφαση αυτή ενός λαού κυρίαρχου που αποφάσισε να ελέγχει, να μην δίνει πια χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας πατριωτισμός οικονομικός, μα απλός πατριωτισμός για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και όλοι πρέπει να πάρουμε παράδειγμα από αυτό. Διάφορα κυκλοφόρησαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πληρώσει ακριβά για να αποθαρρυνθούν άλλοι να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα ή ότι πρέπει να θαυτεί το δημοψήφισμα και το Brexit, να το αγνοήσουμε. Μα δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία του. Τελεία και παύλα. Ποια είναι εναλλακτική ή που θα επιμείνετε στην ε, τεχνοκρατική και ακριβή σας Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζοντας με το πρόγραμμα αυτό που λέει ακόμα περισσότερη Ευρώπη ενώ οι λαοί λένε ότι θέλουν λιγότερη οπότε τότε σας υπόσχομαι ότι πολύ γρήγορα θα καταρρεύσει αυτό το ολοκληρωτικό οικοδόμημα ή που θα βάλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπηρεσία των λαών, στη συνεργασία ελεύθερων εθνών και κυρίαρχων κρατών. Για τη χώρα μου, τη Γαλλία, εγώ αυτό θα κάνω. Θέλω να τη βάλω στο δρόμο της ελευθερίας, που είναι και ο μόνος που οδηγεί στο μεγαλείο. Ζήτω η ελεύθερη λαϊκή έθνη, ζήτω το Ηνωμένο Βασίλειο και ζήτω η Γαλλία. Το λόγο τώρα η κυρία Ντότς ε, από την ομάδα των μη εγγεγραμμένων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου έδωσε την ημιγορία του και την απόφαση αυτή δεν μπορείτε να την αγνοήσετε και ξαναγράψετε. Αναγνώρισαν ότι τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλές ατέλειες και είπαν ας προσπαθήσουμε εμείς να χαράξουμε τη δική μας πορεία. Αυτό το δημοψήφισμα είναι μία νίκη της δημοκρατίας. Δεν είναι το αποτέλεσμα που ήλπιζε ο Πρωθυπουργό μα. Αλλά θα πρέπει να του ε, επενέσουμε που είπαν τη γνώμη του. Για χρόνια ο λαό του Ηνωμένου Βασιλείου προσπαθούσε να σα πει πόσο απογοητευμένο, πόσο ανήσυχο ήταν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί κλείσατε τα αυτιά σα. Αλλά σήμερα ακούτε. Ούτε είναι στιγμή για ψυχραιμία. Αυτοί οι θεσμοί, παρότι άκουσα σήμερα, θα πρέπει να αντισταθούν στο, στη φαγούρα που έχουν για να αντιδράσουν. Το έθνος μας δεν έστρεψε την πλάτη στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Για χρόνια προσπαθήσαμε να έχουμε καλή σχέση με τους Ευρωπαίους ε, συμμάχους. Καλή ε, σχέση. Ε, επιχειρήσεις, ελεύθερο εμπόριο, συνεργασία. Κάτι που θα κάνει τον κόμμα μας πιο ασφαλή, πιο, πιο ευημερή. Αυτό δεν μας κάνει λιγότερο Ευρωπαίους και δεν μας κάνει και λιγότερο αισιόδοξου το Ηνωμένο Βασίλειο όχι μόνο έχει τη δύναμη να τα καταφέρει μόνο του, αλλά επίσης και την εγγενή ανθρωπιά να υπερασπιστεί την ελευθερία των γειτόνων. Ας περιμένουμε με υπομονεσία μια νέα εποχή, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστούν στενά, αλλά ήρεμα για το καλό όλων των λαών. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Γιούγκερ καταρχήν. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής άκουσα πράγματα που ήξερα και πριν από την συζήτηση αυτή. Ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα έθνη στα χέρια των εθνικιστών. Πρέπει να σεβόμαστε τα έθνη, αλλά όχι τους εθνικιστές που δεν είναι πατριώτες, αλλά αντιευρωπαίοι και όχι πατριώτες. Θα ήθελα λοιπόν να πάρουμε τα σωστά μαθήματα από την επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας που πέρασε. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε όλα. Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι η Ευρώπη της λιτότητας. Όλες οι κυβερνήσεις, ακόμα και αυτές που μέσα στην ιστορία ακολούθησαν την ίδια πολιτική. Αυτά που είπε ο κύριος Λάμπερτς δεν τα δέχομαι. Περιέγραψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν να είναι μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή λιτότητας. Εγώ γνώρισα και τους πράσινους και τους οικολόγους όταν ήταν στην κυβέρνηση. Όταν είσαστε στην κυβέρνηση, κάνετε όπω οι άλλοι. Όταν είσαστε στην αντιπολίτευση, εντάξει. Μην δίνετε λοιπόν μαθήματα εσεί στου άλλου, παρακαλώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποφάσισε για τις πολιτικές λιτότητας βάσει αυτών των επιχειρημάτων ή για την προστασία των συνόρων, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στο ευρώ. Άρα οι οικονομικές πολιτικές, οι πολιτικές του ευρώ δεν εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη ζώνη Σέγγεν. Άρα το Ηνωμένο Βασίλειο ελέγχει τα σύνορά του. Συνεπώς μη μας λέτε ότι να είναι. Κύριε Φάρατς, μη μας διηγήσετε ό,τι σας περνάει από το κεφάλι. Πριν από μερικές μέρες παραδεχτήκατε ότι κάνατε λάθος όσον αφορά τα δημοσιονομικά ζητήματα για τη σχέση Συνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το είχατε πει αυτό πριν από το δημοψήφισμα θα σας είχα δώσει συγχαρητήρια. Αλλά είπατε ψέματα. Δεν είπατε την αλήθεια. Μετά αποκαταστήσατε την αλήθεια μετά το δημοψήφισμα. Κύριε Φάρατς, μου αρέσει να συζητάω μαζί σας, γιατί έχουμε και δύο χιούμορ. Και λυπάμαι που είναι η τελευταία φορά που συζητάμε έτσι μεταξύ μας, γιατί είναι η τελευταία φορά που είσαστε εδώ. Πολύ ωραία. Το λόγο λοιπόν έχει εκ μέρους του Συμβουλίου η κυρία Πλασσέρ. Κύριε Πρόεδρε, θα επαναλάβω ότι δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή από το να δεχτούμε και να σεβαστούμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Αυτή λοιπόν τη στιγμή η απάντηση δεν είναι απαραίτητα περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη, αλλά καλύτερη Ευρώπη, πιο πιστική Ευρώπη. Η Ευρώπη των 27 θα συνεχίσει βέβαια να υπάρχει αν αποφασίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να φύγει. Αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Η Ένωσή μας μπορεί να υπάρχει μόνο εφόσον στηρίζεται από τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων και και αν θέλει να τους υπηρετεί και να τους προστατεύει. Αυτή την υποστήριξη δεν πρέπει να τη λαμβάνουμε δεδομένη, πρέπει να εργαστούμε ε, ημέρα και νύχτα όλο το 24 για να το κερδίσουμε. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλες οι απειλές που αντιμετωπίζαμε. Ούτε και όλα αυτά σημαίνουν ότι θα ήταν καλύτερα όλα τα κράτη να λειτουργούν μόνα τους ή απαραίτητα όλοι μαζί συλλογικά. Ξέρετε, οι πολιτικές εξελίξεις υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενότητα καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της ε, τις απειλέ. Γι' αυτό λοιπόν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εργαστούν αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα θέματα που απαιτούν να δραστηριοποιηθούμε. Και ω μια νέα πραγματικότητα ε, τα 27 κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να αποκλίνουν από το να εστιάσουν την προσοχή του στο τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει σήμερα την πραγματικότητα και το μέλλον. Δηλαδή να ασχοληθεί με το προσφυγικό, μεταναστευτικές ροέ να ενισχύσει την ευρωπαϊκή οικονομία δημιουργώντας θέσεις απασχόληση για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ας διασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα διατηρήσουμε τις φιλικές μας σχέσεις σε ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο περίπλοκος. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να απομακρυνθούμε και γι' αυτό ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτόν τον κόσμο τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, δεν αποκλίνουν. Αν κάποιος έχει κουραστεί από αυτή τη συνεργασία, Ας είναι αυτό ένα καμπανάκι όπως λέμε χαρακτηριστικά. Κύριε ε, Πρόεδρε, το ε, Συμβούλιο επιθυμεί να συνεργαστεί όπως πάντα εξάλλου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε τώρα έχει αλλάξει λιγάκι ο κατάλογος των ομιλητών. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ντότς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον τόνο που πήρε αυτή η συζήτηση και ξέρω ότι τα συναισθήματα βράζουν σήμερα το πρωί. Όλα τα στερεότυπα όμως έχουν ενισχυθεί. Τα στερεότυπα τα οποία φοβήθηκαν οι Βρετανοί και καταψήφισαν την Πέμπτη. Δεν θα λειτουργήσουν αυτά, δεν θα πείσουν το Βρετανικό λαό όλα αυτά τα επιχειρήματα. Αυτό που μένει να κάνουμε είναι να αποδεχτούμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, να χτίσουμε σχέσεις που θα είναι αμοιβαίως επωφελείς για όλους τους λαούς η σχέση μας με, σεβα... με σεβασμό των αποφάσεων που θα μας εξασφαλίσει ευημερούσα οικονομία, θα προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα εξασφαλίσει την ειρήνη σε ένα κόσμο ο οποίος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Γιούγκα ε, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από το Κοινοβούλιο που είμαι αναγκασμένος να φύγω. Ο κύριος Τίμερμαν θα μείνει εδώ. Ε, είπε τουλάχιστον ότι με χαρά θα μείνει. Εγώ έχω ένα ραντεβού με τον ε, Βρετανό Πρωθυπουργό και επειδή σέβομαι τη Βρετανική Δημοκρατία είμαι αναγκασμένος να φύγω. Πολύ ωραία κύριε Γιούγκε, Το λόγο λοιπόν έχει ο κύριος Ντεγκράφ. Ευχαριστώ πολύ ιστορικής σημασίας ημερομηνία αυτή της Πέμπτης που μας πέρασε για την ιστορία της Ευρώπης. Η απελευθέρωση από την Ευρώπη άρχισε. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πρώτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει ένα πολύ σημαντικό μέλος της. Είναι η αρχή του τέλους για ένα αποτυχημένο εγχείρημα. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε με τους ψηφοφόρους να υποστήριξε τις ελίτ σε βάρος των λαών της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος σημαίνει ότι πρέπει να επανακτήσουν την κυριαρχία τους οι χώρες, τα κράτη. Και όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κόσμος θέλει να επανακτήσει την κυριαρχία του. Η διαδικασία πρέπει να αρχίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να σταματήσουμε με ε, τη συνέχιση της πορείας αυτής ενοποίησης τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Να επανακτήσουμε τα σύνορά μα. Το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό δήλωσε ότι θέλει τα δικά του, τα σύνορα, τη δικιά του πολιτική, τη δική του κυριαρχία. Απελευθέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ολλανδία, την Ρουμανία και άλλες χώρες αυτό ακριβώ ισχύει. Και είπε ο κύριο Γιούγκερ, μα σταματήστε. Αποτύχατε κύριε Γιούγκερ για να τα καταφέρετε. Σταματήστε κύριε Γιούγκερ και οι υπόλοιποι επίτροποι, η νέα επιτροπή στην ίδια αυτή πορεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάραντς τώρα έχει το λόγο εκ μέρους του FDD. Σήμερα το πρωί οι χρηματαγορές αυξήθηκαν. 12% αυξήθηκαν. Είναι αδύναμη η στερλίνα, αλλά ούτως ή άλλως από τον Ιούλιο του 2014 άρχισε να πέφτει. Και οι πρόεδροι τώρα τη ε, Νέα Ζηλανδία ε, και τη Αυστραλία ε, μπαίνουν στη σειρά για το ποια θα είναι η πρώτη χώρα που θα κάνει business που θα κάνει εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλά είναι τα πράγματα. Η μόνη, το μόνο πρόβλημα αναταράξει και τα λοιπά είναι οι πολιτικέ αναταράξει. Ε, παρετήθηκε ο Λόρτο Χιλ. Ο... Παρετήθηκε ο Πρωθυπουργό, λέει ο κύριο Φάρατ. Υπάρχει αυτή ανατα... η αναταραχή στην πολιτική που μπορεί όμω να είναι και πολύ καλό πράγμα, πολύ υγιέ πράγμα. Εγώ μπήκα στην πολιτική γιατί η πολιτική μα στην Ευρώπη ε, μας οδήγησαν στο ευρωπαϊκό πολιτικό project. Ελπίζω λοιπόν ε, τα αποτελέσματα της περασμένης εβδομάδας να παρασύρουν ε, μερικούς από αυτούς τόσο το καλύτερο. Το λόγο έχει ε, επόμενο ομιλητή, ο κύριο Σμιτ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ εκπροσωπώ τη Σκοτία και πρέπει να σας πω ότι είμαι υπερήφανος Σκοτσέζος αλλά είμαι και υπερήφανος Ευρωπαίος. Θέλω η χώρα μου να είναι ανοιχτή, διεθνιστική ας το πούμε, δίκαιη, ευρωπαϊκή, με οικολογική στάση και οι κάτοικοι της Σκοτίας μαζί με αυτούς της Βόρειας Ιρλανδίας ε, και του Λονδίνου και του Σουαλίας και της Αγγλίας, ε, πολλοί λοιπόν και περισσότεροι εξ αυτών αποφάσισαν να παραμείνουν σε αυτή την οικογένεια κρατών. Ε, σας το υπενθυμίζω λοιπόν αυτό και είναι κάτι που πρέπει να γίνω σεβαστό. Συνάδελφοι, υπάρχουν πολλά που θα είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πρέπει να παραμείνουμε νυφάλοι, αλλά μην ξεχνάτε ποτέ αυτό η σκοτία δεν σας εγκατέλειψε, δεν σας πρόδεσε. Σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, μη μας εγκαταλείψετε και μας τώρα αυτή τη στιγμή. Εκ μέρους της Ενωμένης Αριστεράς, το λόγο έχει η κυρία Άντερσον. Οι ευρωβουλευτές όπως η Νταϊάν Ντότζ, η Μάριν Λεπέν, θα έλεγαν ότι εμείς στη Βόρεια Ιρλανδία είμαστε δεσμευμένοι από την ε, Βρετανική ψήφο. Εμείς λέμε όχι, δεν είμαστε. Και όπως και ο προηγούμενος ε, Ευρωβουλευτής, ο κύριος Σμιθ, σας ζητάμε να σεβαστείτε τη δική μας ψήφο. Την υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε την ψήφο του λαού της ε, Βόρειας Ιρλανδίας, όπως και οι Σκοτσέζοι το ίδιο, που ψήφισαν υπέρ της παραμονής. Δεχόμαστε, σεβόμαστε. Σεβόμαστε και δεχόμαστε και υπερασπιζόμαστε τη θέληση του λαού της Βόρειας Ιρλανδίας. Αν όμως η αγγλική ψήφος μας οδηγήσει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σαν να αποφασίζει η Βρυτάνια. Έγινε δημοκρατική ψηφοφορία. Ψηφίσαμε να παραμείνουμε. Σας λέω ότι το τελευταίο πράγμα που ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας χρειάζεται είναι σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύνορα με τα 27 κράτη-μέλη και πού θα σταματάνε αυτά τα σύνορα, στη μέση της Ιρλανδίας. Εσείς υποστηρίξατε την ειρηνευτική μας διαδικασία. Σας ζητάω να συνεχίσετε να κάνετε ακριβώς αυτό. Το Sinn Féin, εμείς δουλέψαμε για να υπάρξει μια ισχυρή ψήφο υπέρ τη παραμονή. Για περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη κοινωνική Ευρώπη, πιο δημοκρατική Ευρώπη. Και το λέω στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Δεν ακούτε. Δεν συνειδητοποίησατε το μέγεθος της αντιπολίτευσης του, των απλών λαών. Δεν συνειδητοποίησατε τις αντιδημοκρατικές πρακτικές και τις αντικοινωνικές πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές θα πρέπει να αλλάξουν. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιβιώσει, πρέπει να τα ακούσετε όλα αυτά. Σας ζητάω όμως να σεβαστείτε την ψήφο του λαού της Βόρειας Ιρλανδίας. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Εκ μέρους των ε, φιλελευθέρων, ο κύριος ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, ε, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνοντα αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όσου παρίστανται εδώ και να εκπέμψουμε τώρα όλοι μα ένα χειρό μήνυμα προ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι όλοι μας μαζικά να υπερψηφίσουμε το ψήφισμα το οποίο έχουμε προετοιμάσει για αυτή την Ολομέλεια. Και να μην αρχίσουμε τώρα να λέμε «Α, δεν μου αρέσει το Α ή το Β». Αυτό που έχει τώρα πολιτική σημασία είναι μαζική υπερψήφιση του δημοψηφίσματος. Και το τελευταίο που θέλω να πω, απευθύνομαι προς τον κύριο Φάρατς. Κύριε Φάρατς, έχω σοκαριστεί. Εσείς παρουσιάζεστε εδώ ως ο αμύντορας του απλού μέσου ανθρώπου, του σκληρά εργαζόμενου και εσείς έχετε μία offshore εταιρεία εξωχώρια εταιρεία οικοδομικών και ε, κατασκευών. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει για το μέσο άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει. Ε, θα πρέπει κάπως να δούμε λιγάκι και το θέμα της, ε, του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μην ξεχνάτε 70 ολόκληρα χρόνια με συγχωρείτε, 17 ολόκληρα χρόνια πληρώνουμε το μισθό σα. 17 ολόκληρα χρόνια σας πληρώνουμε ως Ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Λεγκούτκο. Πρέπει να σας πω πως έχω απογοητευτεί κάπως από τη συζήτηση αυτή. Έχει συμβεί κάτι πολύ κακό στη συζήτηση για το Brexit. Εντάξει, μπορεί να είναι κακό, επικίνδυνο, όχι όμως για το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο μια χαρά θα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι κακό και επικίνδυνο συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το χειρότερο που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τι κάνετε εσείς ξανά και ξανά επανέρχεσαι στις ίδιες ρυθμίσεις, λέτε τα ίδια και τα ίδια, είναι τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιες προσβολές, ξανά και ξανά με συναισθηματισμούς και εξάρσεις. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε ότι οι ηγέτες μας κάνανε κάτι πολύ κακό. Η Επιτροπή λοιπόν τι θα κάνει για να διορθώσει τα πράγματα. Η πλειοψηφία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να κάνετε κάτι διαφορετικό. Εν εσείς παίζετε συνέχεια το ίδιο σκοπό. Τα βάζετε με τους σοβινιστές. Δεν έχετε δηλαδή τελικά καταλάβει ποια είναι η πραγματικότητα της σήμερον ημέρα, το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς συνεχίζετε με τον ίδιο σκοπό. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τα πράγματα φυσικά δεν είναι ρόδινα Είμαστε ένα ζωντανό οργανισμό που μπορεί να μάθει από τα σφάλματά του. Εμεί συμφωνούμε γι' αυτό. Ελπίζω και οι υπόλοιποι ηγέτε να συμφωνούν επίση. Από τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Ένα πράγμα στον κύριο Φάρατζ. Εγώ δεν σφυρίζω. Δεν αποδοκιμάζω σφυρίζοντα. Ακόμα και αν ήξερα να σφυρίζω όμω, δεν θα το έκανα ποτέ απέναντι στου συναδέλφου. Και για κανέναν θα το έκανα. Ένα πράγμα να σα πω, κύριε Φάραντζ. Εσεί δεν κάνετε καλό στη χώρα σα. Και η ιστορία θα το αποδείξει. Δυστυχώ η ιστορία θα το δείξει αυτό. Και θα το αποδείξει. Δεν είναι στιγμή τώρα για να πολεμούμε ο ένας τον άλλον. Για να χειραγωγούμε. Είναι μια σημαντική ιστορική στιγμή. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αν θέλανε κάποιοι τον Brexit, να το. Και τώρα δεν καταλαβαίνουμε γιατί καθυστερείται. Τι λέει η δημοκρατία. Θα πρέπει να καταγράψετε ποιο είναι το αποτέλεσμα και να προχωρήσετε στην επόμενη κίνηση. Να πάτε στην κοινοποίηση. Δεν μπορούμε να αφαιθούμε, ας πούμε, στις εσωτερικές, ε, στα εσωτερικά μαγειρέματα και στα παιχνίδια του συντηρητικού κόμματο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να περιμένουμε τι θα πει το συνέδριο των Τόρι. Αυτό είναι απίστευτο, είναι παράλογο. θα πρέπει να ε, εξεγερθούν αυτό το 52% των Βρετανών που ψήφισαν υπέρ του Brexit με αυτέ τι καθυστερήσει. Είναι σαφέ τώρα ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να υποφελθούν από αυτή την ψήφο για να καταστρέψουν. Εμεί είμαστε στην αντίθετη όχθη και έχουμε καλή παρέα εδώ. Έχουμε του χριστιανοδημοκράτε, έχουμε του φιλελεύθερου, έχουμε του πράσινου. Έχουμε όλου όσου θέλουν να αλλάξουν και να σώσουν την Ευρώπη. Είπαμε ότι πρέπει να γίνει πάρα αυτά μάλιστα. Και ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μας λάβει υπόψη, να λάβει υπόψη το αίτημά μας. Αλλά κοιτάμε και προς το μέλλον. Και το βραχυπρόθεσμο και το μεσοπρόθεσμο. Σκεφτόμαστε μία συνέλευση ανοιχτή στους πολίτες. Με τους πολίτες. Όχι, τις ελίτ, όχι μόνο με τις ελίτ των Βρυξελών. Ούτως ώστε να φτιάξουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για μία διαδικασία πολιτικής ολοκλήρωσης πιο έντονης. Που θα προβλέψει και έναν Υπουργό ε, Οικονομικών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα καλύτερο προπολογισμό, κοινέ πολιτικέ άμυνα, ε, καταπολέμηση τρομοκρατία, ε, ένα ευρωπαϊκό FBI, κοινέ πολιτικέ για τη μετανάστευση. Για τη μετανάστευση. Αυτά είναι τα δικά μα θέματα που θέλουμε να προχωρήσουμε, να τα προωθήσουμε πολύ γρήγορα και μεσοπρόθεσμα. Και τα θέλουμε να τα κάνουμε αυτά ενωμένοι, ξεπερνώντα τι διαφορέ μα που παραμένουν αλλά που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μπουν λίγο στην άκρη σε αυτή την κοινή προσπάθεια για να διασώσουμε την Ευρώπη. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτή θα την προωθήσουμε και μάλιστα με μεγάλη στεναρότητα. Εκ μέρου του ΕΛΚ, για άλλη μια φορά, το λόγο έχει ο κύριο Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι σήμερα είχαμε μια ιδιαίτερα καλή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ε, κατέστη σαφές ε, πρώτον του τι, το τι είδους ε, προκλήσεις αντιμετωπίζουμε. Δεν αξίζει καν τον κόπο να σχολιάσει κανείς αυτά που λέει ο κ. Φάρατζ γιατί πού να ξέρουμε μετά από δύο εβδομάδες μπορεί να ισχυρίζεται άλλα. Δεν σχολιάζω λοιπόν. Και για την κυρία Λεπέ να πω η κυρία Λεπέν κατέστησε απόλυτα σαφές ότι κατ' ουσίαν δεν έχει καμία απάντηση να δώσει στην ασάφεια και ανασφάλεια των, των Βρετανών. Και οι Βρετανοί θέλουν να πιστεύουν ότι οι Βρετανοί έχουν πρόβλημα και ότι δεν έχει ίδια. Μα δεν είναι αλήθεια. Αυτά δεν είναι πιστικά επιχειρήματα. Αυτά τέλος πάντων ήταν ένα κομμάτι της συζήτησης. Το δεύτερο όμως πιο σημαντικό είναι ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταστήσαμε σαφές ότι εμείς στηρίζουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα, επιθυμούμε να προχωρήσουμε και παρακαλούμε, ειλικρινά παρακαλούμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί να μην προ προχωρήσει σε αντιπαραθέσεις. Αυτό το ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Να μην τσακώνονται, αλλά να δείξουν όλοι ότι πιστεύουν σε αυτή την Ευρώπη και επιθυμούν να την οικοδομήσουν περαιτέρω. Πρόεδρος, ε, τελείωσε.